Ladies gentlemen, good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορούμε μήπως να αρχίσουμε. Mm-hmm. Έχω μια ανακοίνωση. Δηλαδή ότι χρειάζεστε τις κάρτες για την ψηφοφορία. Παρακαλώ λοιπόν βγάλτε τις. Ετοιμάστε τις. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω τώρα για τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Για τον ορισμό εισηγητών, ο κύριος Μαρίνου Επίντου ορίστηκε εισηγητής για την άρση της ασυλίας του Νταν Νίκα. Ο Αντρέι Ντούντα για την άρση της ασυλίας του Σεργέη Στάνισεφ, η κυρία Χάουταλα για την άρση της ασυλίας του Ζερόμ Λαβριέ και για τους υπόλοιπους ηγητές για το νομικό υπόβαθρο κυρία Χάουταλα για την επικουρικότητα η κυρία Φεράρα για διαφορές ο κύριος Καβαντά για την επιτροπολογία και λοιπά. Ο κύριος Σάγερ για κωδικοποιήσεις και recast. Ο κύριος, η κυρία Μαστάλκα συντάκτες ονομοδοτήσεων. Αποφασίστηκε η διάμεση έκθεση για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα Accountability and integrity in the EU. στους σοσιαλιστές και για τη διαφάνεια από τον πρόεδρο. Για τα ψηφίσματα οι συντονιστές αποφάσισαν Χρωμοδότηση με μορφή επιστολής σύμφωνα με το 133 του κανονισμού για το ψήφισμα της κυρίας Μπιζότο για την 3η Νοεμβρίου για την ε, μάλλον ασυμβατότητα του Δημοσιονομικού Συμφώνου με τη συνθήκη της Λισαβόνας και οι συντονιστές σημείωσαν ότι υπάρχει ψήφισμα του Άλντο Πατρίτσελο για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Υιοθεσιών. Επίσης συμφώνησαν οι συντονιστές να ζητήσουν επίσκεψη της Επιτροπής μας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο το δεύτερο μισό του 2015 κατόπιν ετήσεως από τον πρόεδρό του Μπενουά Μπατιστέλη. Οι συντονιστές συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας για νομικά θέματα που αφορούν την ρομποτική. Η συγητής ορίστηκε η κυρία Ντελβό. Αποφάσισαν επίσης ένα μέλος της ΙΝΤΑ και ένα μέλος της γραμματείας της να προσκληθούν στις εργασίες της ομάδας εργασίας για τα πνευματικά δικαιώματα ανάλογα να προσκαλούνται ανάλογα με το θέμα κάθε φορά. Συμφώνησαν να ζητήσουν από το τμήμα χάραξης πολιτικής να κάνει προτάσεις νομικής εμπειρογνωμοσύνης στην Ένωση. και το χρονοδιάγραμμα επισκέψεων του 15 εγκρίθηκε επίσης από τους, εισηγητάς, από τους συντονιστάς. Επίσκεψη στη Λετωνία με άγνωστες ακόμα ημερομηνίες. Στην Ελλάδα 18 με 20 Μαρτίου. Στη Σουηδία 8 με 10 Απριλίου. Ουάσιγκτον 8 με 10 Απριλίου επίσης, Χάγη 5 Μαΐου και Κίεβο 18 και 19 Ιουνίου. Η νομική υπηρεσία θα κάνει μια παρουσίαση γνωμοδότησης για, με θέματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τη δημιουργία μιας συνθήκης για ένταξη της Ένωσης στην υπάτη ε, ε, αρμοστία, στην ΕΣΦΑ. Οι επιτροπές Τραν και Ήτρε During the committee. θα συμφωνήσουν για το καλοκαίρι. Θερινή ώρα, για τη θερινή ώρα θα συμφωνήσουν. Την τρίτη όμως ή την πέμπτη αντί το απόγευμα της Τετάρτης. Αυτές είναι οι αποφάσεις των συντονιστών και συντονιστριών. Και τώρα πάμε στο σημείο 12. Σημεία 12 με 19 επιτρέψτε μου. Και εάν η κυρία Χάουταλα θέλει να πάρει το λόγο, θα την παρακαλούσα διότι είναι η για τα σημεία αυτά. Αλλιώς προτείνω να ψηφίσουμε μαζί από κοινού το σύνολο αυτών ε, των προτάσεων. Κυρία Χάουταλα πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. προτείνω να ψηφίσουμε τώρα και να μην τροποποιήσουμε τις εκθέσεις, διότι το Συμβούλιο είχε πολύ χρόνο για να συμφωνήσει και γι' αυτό δεν συμφωνώ και με την τροπολογία για παράταση του χρόνου. Να δώσουμε παράταση δύο μηνών, δηλαδή από δύο σε τέσσερις μήνες. Και να προσθέσω κάτι που νομίζω ότι θα αναφέρει και η κυρία Χάνιπολ. Είχαμε συζητήσεις σχετικά με το δυναμικό των 8 τρίτων χωρών, σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις ε, συμβάσεις της Χάγης. Και νομίζω ότι η κυρία Χάνιπολ θα αναφερθεί στο θέμα αυτό. Κατά τα άλλα, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε στη ψήφο, στην ψηφοφορία. Κυρία Χάνιπολ, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Αλλά με απασχολούν τα οχτώ αυτά κράτη και το κατά πόσο είναι κάποια από αυτά σε θέση να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις τη Σύμβαση της Χάγης. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, τα κράτη-μέλη ζήτησαν αξιολόγηση των κρατών με τα οποία πρόκειτο να συνάψουν ε, συμφωνίες. Ε, και τώρα αυτή η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γίνει κάτι όμως όσον αφορά αυτές τις αξιολογήσεις. Ωστόσο, καταλαβαίνω επίσης ότι κάποιες από αυτές τις χώρες δεν έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες διαδικασίες. Τα περισσότερα κράτη όμως καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες. Το Ευρωπαϊκό Νομικό Ινστιτούτο και άλλοι θεωρούν ότι ο καλύτερος τρόπος να τα καταφέρουν οι χώρες αυτές είναι να προσχωρήσουν στη σύμβαση. Γι' αυτό δεν είμαι κατά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπερψηφίσουμε τις προτάσεις αυτές, θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε την κατάσταση στις χώρες για τις οποίες μιλάμε. Και γι' αυτό προτείνω να πραγματοποιηθεί ακρόαση για το θέμα αυτό στο εγγύς μέλλον για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πιο αναλυτικά τις λεπτομέρειες και να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. Επίσης, προτείνω κατά την επίσκεψή μας στην Χάγη να εξετάσουμε τη σύμβαση αυτή επί τόπου. Thank you very much. Uh, we can Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτα θα ψηφίσουμε πάνω σε 8 όμοιες τροπολογίες του κυρίου Τζαμπάσκη. Σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Από ό,τι κατάλαβα, η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ? Ποιος είναι κατά? Αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ψηφίσουμε με τις ηλεκτρονικές κάρτες. Ψηφίζουμε το σύνολο των σχεδίων εκθέσεων. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Uh, One too many EPP and one too many ALDE voting. Uh -huh. I have the information that there are too many people voting. Ψήφισαν υπερβολικά πολύ. Δύο παραπάνω από το ΕΛΚ από ό,τι θα έπρεπε και ένας παραπάνω από την ΑΛΔΕ. Ενδιαφέρον. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η τροπολογία. συγγνώμη, εγκρίθηκαν τα σχέδια εκθέσεων. Θα ξαναψηφίσουμε για το σχέδιο νομοθετικών ψηφισμάτων. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. Συγχαρητήρια κυρία Χάουταλα. Προχωράμε στο σημείο 20. προώθηση της ελεύθερης κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων. Δίνω το λόγο στην κυρία Ντελβό που είναι η συγγήτρια. Συγγνώμη. Έχω μπερδευτεί, διότι νόμιζα ότι επρόκειτο να ψηφίσουμε την εντολή διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Πρόεδρο, εάν δεν χρειάζεται να σχολιάσετε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Σημείο 21. πιστοποίηση δεξιοτήτων και θα ήθελα να πω ότι από το σχέδιο έκθεσης έχουν αποσυρθεί κάποιες τροπολογίες. Αναφέρεται αυτό στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε σηκώνοντα τα χέρια. Και η τελική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Παράγραφος 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές έχουμε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού 9 έως 15 τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατόπιν έχουμε μία προφορική τροπολογία. Η εντολή του κυρίου Φίλιπ Μπράτπορν έληξε στις 21 Δεκεμβρίου του 2014. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα συγχαρώ τον εαυτό μου λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. 22, 22. Να ψηφίσουμε κατευθείαν. Ποιος είναι υπέρ. Διανάταση χειρός. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προχωράμε τώρα στο σημείο 23. Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών. Το λόγο τον έχει η κυρία Γκέριγκερ. Συγχωρείτε, ο κύριος Ντούντα ζητάει το λόγο επί της διαδικασίας. Ε, ευχαριστώ. Ναι. Επί της διαδικασίας έχω ένα αίτημα, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να παρακαλέσω μετά την ψηφοφορία το σημείο 34 να αναβληθεί. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Yes, I think that is, that is viable. Ναι, νομίζω ότι γίνεται. Ε, ή μπορούμε να το κάνουμε ως το τελευταίο σημείο του πρωινού πριν το μεσημεριανό διάλειμμα. Συμφωνείτε? Uh, Yes, yes, yes. Ναι, ναι, ναι, βεβαίω. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Γκέριγκερ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Για το κανονισμό της επίλυσης μικροδιαφορών. 86 τροπολογίες κατατέθηκαν, ευχαριστώ τους συντάκτες τους. Πολλές τροπολογίες, πολλές, συμπληρώνουν και βελτιώνουν το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Λοιπόν, πρώτα πρώτα. Από πού προέρχεται αυτή η πρόταση νέου κανονισμού γενικά. Η Κομισιόν αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα διαδικαστικά για την επίλυση μικροδιαφορών και ότι τα προβλήματα αυτά τίθενται για μικρά ε, ποσά άρα για διαμεθοριακές κυρίως διαφορές εδώ το πρόβλημα είναι η έλλειψη πληροφόρησης γιατί καμιά φορά δεν γνωρίζει κανείς τι νόμοι ισχύουν σε τρίτες χώρες και πώς λειτουργούν τα δικαστήριά τους. Χρειάζεται μετάφραση, διερμηνία, επιτόπια επίσκεψη κτλ. Όλο και περισσότερες διαμεθοριακές διαφορές σημειώνονται και έπρεπε επομένω να βρεθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης τους για να λειτουργεί καλά η οικονομία. Με μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν είδα αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Κατέθεσα βέβαια και οι ίδια μερικές τροπολογίες, αλλά γενικά η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή και σωστή. Θα ήθελα η διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη για την χρήση από τους πολίτες όπου και να βρίσκονται και όποια γλώσσα και να μιλάνε. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 11 τονίζει ότι η συχνότητα της προσφυγής στα δικαστήρια για μικροδιαφορές στα κράτη-μέλη είναι πολύ χαμηλή. Γι' αυτό χρειάστηκε απλοποίηση για την επίλυση και διαμεθοριακός. Πρώτα βέβαια έπρεπε να οριστεί τι είναι μικροδιαφορά και συμφωνώ από αυτού με την πρόταση της Κομισιόν που λέει, που λέει ότι για τις διαμεθοριακές δοσοληψίες θα θεωρούμε μικροδιαφορά μέχρι 10.000 ευρώ. Το τωρινό όριο είναι 2.000 ευρώ και έτσι δεν θα επέτρεπε την εφαρμογή αυτού του κανονισμού γιατί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες διαφορές αφορούν ποσά πάνω των 10.000 ευρώ. Για να διευκολυνθούν λοιπόν οι δραστηριότητες τους ιδιαίτερα οι διαμεθοριακές των δοσοληψίες είναι καλό το όριο να μπει στα 10.000 ευρώ είναι εύλογο και θα λύσει πολλά προβλήματα ακόμη κάτι πολύ συχνά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοούμε μικροδιαφορές ο όρος αυτός μπορεί να οδηγήσει μερικούς σε παρεξηγήσεις γιατί μια μικροδιαφορά ορίζεται ανάλογα με το μέσο εισόδημα. Για μερικές χώρες 10.000 ευρώ μπορεί να θεωρείται κολοσιαίο ποσό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματος χάρη τα small claims, οι μικροδιαφορές, θεωρούνται μέχρι 12.000 θερλίνες. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί του τι είναι μικροδιαφορά. Και για να μην υπάρχουν λοιπόν παρεξηγήσεις πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος αυτός με τον όρο διαφορά μέχρι 10.000 ευρώ. Μπορεί κανείς να μιλήσει για απλοποιημένη διαδικασία για επίλυση διαφορών μέχρι 10.000 ευρώ. Έτσι μόνο θα υπάρξει αποτέλεσμα διότι όπως σας είπα πριν δεν αφορά μόνο τους απλούς πολίτες, πρέπει όλοι, οι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γνωρίζουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Η τροπολογία 30, τροπολογία 30 λέγω, στοχεύει στην τροποποίηση του ορίου για ιδιώτες, ένα ανώτατο όριο διαφορετικό για τους ιδιώτες από ό,τι για τις επιχειρήσεις. Αυτό μπορούμε να το ξανασκεφτούμε. Αλλά νομίζω ότι θα καταστήσει τα πράγματα πιο δύσκολα. Πρέπει οι κανόνες να είναι διαφανείς, απλοί και εύληπτοι για όλους. Και για τους ιδιώτες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα για το όριο των δικαστικών εξόδων. Και αυτό έχει συζητηθεί πολύ. Εδώ δεν καθορίζουμε όρια γι' αυτό. Διότι το θέμα αφορά καθαρά τα κράτη-μέλη και τον τρόπο λειτουργίας του δικαστικού των συστήματος. Θέλουμε απλώς τα δικαστικά έξοδα να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα και να ανταποκρίνονται να μην είναι δυσανάλογα με το ποσό που εκδικάζεται. Αν τα δικαστικά έξοδα είναι παραπάνω από ότι το, η διαφορά, ε, τότε δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε. Γιατί έτσι θα οδηγηθούμε σε περισσότερη ατιμορρησία και παρανομία. Υπάρχει επίσης το θέμα των ελαχίστων δικαστικών εξόδων για να αποφεύγεται, να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των περιπτώσεων, των υποθέσεων για χαμηλά ποσά. Ας πούμε ελάχιστα δικαστικά έξοδα 34 ευρώ. Ναι, να μην υπάρχουν χαμηλότερα από 34 ευρώ δικαστικά έξοδα. Χαίρομαι γιατί όλοι υποστηρίξατε την πρόταση δυνατότητας πληρωμής με πιστοτική κάρτα ή με έμβασμα γιατί αλλιώς έπρεπε να πάει κανείς από το προσώπο στο δικαστήριο να πληρώσει. <clears throat> Τώρα υπάρχει νέα δυνατότητα <clears throat> να πληρώνονται τα δικαστικά έξοδα όπως σας είπα και χαίρομαι γιατί και το Συμβούλιο δεν αντιτάχθηκε. Δεν αντιτάχθηκε. Μερικές τροπολογίες επιτρέπουν την συμπλήρωση και βελτίωση της αρχικής πρότασης της Κομισιόν όπως η 72 που προτείνει τα δικαστικά έξοδα τα δικαστικά έξοδα να μην ξεπερνούν εκείνα που θα ζητιούνταν από ανάλογη περίπτωση αν δεν χρησιμοποιούνταν η απλοποιημένη ευρωπαϊκή διαδικασία. Ούτε να αυξάνονται τα δικαστικά έξοδα αν η περίπτωση είναι διαμεθοριακή. Πολύ καλή πρόταση αυτή, θα την υποστηρίξω. Υπάρχουν και άλλες καλές τροπολογίες που αφορούν, που αφορούν τις υπηρεσίες παραδείγματος χάρη την βοήθεια συμπλήρωσης εγγράφων, πολύ καλή τροπολογία. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα περάσει, θα γίνει δεκτή από το Συμβούλιο, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες για την εφαρμογή των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας που προβλέπει ο κανονισμός. Εδώ πρέπει να βρεθεί ένας σωστό συμβιβασμός. Όλοι ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους κάποια προθεσμία μέχρι να μπορέσουν να εφαρμόσουν κάποια μεταβατική περίοδο τον νέο αυτό κανονισμό. Μπορεί μερικές περιπτώσεις να μπορούν να λυθούν με τηλεδιάσκεψη. Αλλά γι' αυτό απαιτείται να έχουν εγκαταστάσει στα δικαστήρια που δεν τα ε, έχουν όλα ακόμα. Να αυτά είχα να σας πω για τις τροπολογίες και αναμένω τώρα τα σχόλιά σας. Θα συνεχίσουμε την εργασία για την επίτευξη ικανοποιητικού συμβιβασμού για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα ώστε να αποτελέσει μία από τις επιτυχίες της Λετωνικής Προεδρίας. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. Κύριε Χάνιμπολ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και συμφωνώ με όσα είπε. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ αφορά το ζήτημα της ενημέρωσης γιατί η διαδικασία αυτή δεν έχει υιοθετηθεί ε, ευρέως γιατί ο κόσμος δεν την γνωρίζει. Οπότε, όταν μιλάμε για αυτό το θέμα, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τρόπους ενημέρωσης ε, του κοινού. Ευχαριστώ. Κύριος Ράντιεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει και να πω πως η διάκριση του κατοφλίου για φυσικά και νομικά πρόσωπα αντιστοίχως νομίζω πως συμβαδίζει με την οικονομική πραγματικότητα το να βάλουμε το κατόφλι πάνω από τα 10.000 ευρώ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο δεδομένου του ότι μιλάμε για μικροδιαφορές ε, ούτως ή άλλως και επιπλέον θα πρέπει νομίζω να μην ε, δώσουμε περαιτέρω αρμοδιότητες ε, στα δικαστήρια για μικροδιαφορές που μπορούν να πάνε άνετα στα εθνικά δικαστήρια. Αν λοιπόν μιλάμε για διαφορές εντός ενός κράτους μέλους, εκεί πέρα πρέπει να γίνει και η εκδίκαση για να μην διαλέγει κανείς ε, το που θα πάει. Όσον αφορά τώρα την ε, τηλεδιάσκεψη, όταν κάποιος διάδικος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, τότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα της ε, τηλεδιάσκεψης και πρέπει να ενθαρρύνουμε τα δικαστήρια να έχουν τον αναγκαίο εξοπλισμό. Ε, γι' αυτό ακριβώς πρέπει νομίζω να δοθεί αυτή η προθεσμία των δύο ετών για να μπορέσουν να εξοπλιστούν τα δικαστήρια. Κύριε Μπουντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της. Νομίζω πως είναι απολύτως απαραίτητο και είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει το κοινό γιατί θα είναι ένα στοιχείο χρήσιμο για όσους έχουν μικροδιαφορές στα κράτη-μέλη. και βεβαίως θα ισχύει μόνο όταν υπάρχει ακριβώς ένα διεθνές στοιχείο στην υπόθεση. Όχι αν πρόκειται για μια καθαρά εθνική ε, υπόθεση. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να τονίσω το εξή, θα ήθελα να επιμείνω στην διαφοροποίηση για το πλαφών ε, για τα νομικά πρόσωπα και τα πρόσωπα που εξομοιώνονται με αυτά γιατί βεβαίως η οικονομική της δραστηριότητα είναι υψηλότερη από αυτή των φυσικών ε, προσώπων. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο θα είναι στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν αυτές έχουν προβλήματα. Επιπλέον, καλό είναι να μην μένουμε μόνο ε, στο τι μπορεί να γίνει εκ αλλά και στα προληπτικά μέσα γιατί αν μια εταιρεία ε, σκεφτεί ότι υπάρχει δυνατότητα να μην πληρώσει τα χρέη θα το ξανασκεφτεί όταν ξέρει ότι υπάρχει κάποιο μέσο τέτοιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολο. Βεβαίω θα είναι συλλογική η απόφαση. Είναι δύσκολο να αποφασίσουμε το τι είναι μικροδιαφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Ρουμανία ή σε άλλο κράτος μέλος. Αλλά εάν σκεφτούμε το ποσό των 10-15 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για μια μεταφορική εταιρεία είναι δύο-τρεις διαδρομές από τη μια άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη. Τώρα όσον αφορά την προθεσμία για την εφαρμογή στα κράτη-μέλη νομίζω πως μια λογική προθεσμία είναι οι 12 μήνες. Ε, οι 6 μήνες δεν είναι ρεαλιστική γιατί δεν μπορεί να οργανωθεί ο πληστηριασμός για τον εξοπλισμό πληροφορικής. 12 μήνες νομίζω είναι καλύτερη η προθεσμία για την εφαρμογή του κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σουσπάσκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις τροπολογίες που συζητάμε τώρα. Υποστηρίζω τις τροπολογίες που καθορίζουν σαφώς τις διαφορές μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων. Και τώρα είναι σαφές πως η διαδικασία αυτή θα αφορά όχι μόνο τις εταιρείες αλλά όλους τους πολίτες της Ένωσης. Οι τροπολογίες που αφορούν το όριο επίσης ε, εκεί πέρα εντάσσονται. Θεωρώ λοιπόν πως θα ήταν χρήσιμο να έχουμε διαφορετικά κατόφλια για τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα. Η πρότασή μου είναι να μείνουμε στα 10.000 για τα νομικά πρόσωπα και 4-5.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και κάποιες άλλες ε, τροπολογίες αφορούν το είδος ε, των ε, διαφορών. Είτε μιλάμε για όλες τις διαφορές, διεθνείς ή όχι, είτε μιλάμε για τις διαφορές οποίες, οι οποίες έχουν ένα διασυνοριακό στοιχείο. Νομίζω λοιπόν πως θα ήταν χρήσιμο η διαδικασία αυτή να εφαρμοστεί ε, όσο δυνατόν πιο ευρέως. Γιατί θα είναι έτσι η κατάσταση απλούστερη, γρηγορότερη και πιο φτηνή από όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που προτείνονται ε, στα εθνικά δικαστήρια. Οπότε δεν στηρίζω τους περιορισμούς που προτείνονται Θα ήθελα να υποστηρίξω την χρήση ηλεκτρονικών μέσων όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση τους. Όσον αφορά τώρα το τι θα κοστίζει αυτό. Νομίζω πως θα μας δοθεί τώρα μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τα δικαστήριά μας στον 21ο αιώνα. Οπότε νομίζω ότι και οι προθεσμίες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σφιχτές για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή έκθεση που μας παρουσίασε. Τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Καταρχάς συμφωνώ με την κυρία Χάνιμπολ Πολύ συχνά δεν χρησιμοποιείται αυτή η διαδικασία λόγω έλλειψης γνώσης για τη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να εφαρμόσουμε μέτρα για να γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα τη διαδικασία αυτή. Τι είναι μια μικροδιαφορά. Εκτιμώ ότι αναφερθήκατε στη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ότι μια μικροδιαφορά είναι κάτω των 12.000 ε, λιρών. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις από 3.500 ευρώ μέχρι τα επίπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο τρόπος που ορίζεται η μικροδιαφορά εξαρτάται από την οικονομία και από το μέσο εισόδημα. Εάν εξετάσουμε λοιπόν τις μέσες μηνιές αποδοχές στα κράτη-μέλη, κυμαίνονται από κάποιες εκατοντάδες ευρώ μέχρι περίπου 2.000 ευρώ. Εάν λοιπόν παρουσιάσουμε μία διαδικασία η οποία να ισχύει για εταιρείε περιορισμένη ευθύνη αλλά και για φυσικά πρόσωπα, χωρί περιορισμένη ευθύνη αλλά και με πιο περιορισμένου πόρου, θα πρέπει να γνωρίζουμε το κοινωνικο-οικονομικό σενάριο στο οποίο κινούμαστε. Συμφωνώ λοιπόν με τη διάκριση ανάμεσα στα φυσικά πρόσωπα και στα νομικά πρόσωπα όσον αφορά το όριο. Η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά μέσα για τη συλλογή πληροφοριών, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό είναι κάτι που αφορά κάθε νομικό σύστημα. Να γνωρίζω όμως ότι όχι όλα τα κράτη-μέλη ότι δεν έχουν εισάγει όλα τα κράτη-μέλη επαρκή πόρους για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και γι' αυτό θα πρότεινα 12 μήνη προθεσμία αντί για εξάμηνη για την εφαρμογή της οδηγίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πως ε, είμαι θετικός ως ε, προς αυτό το σύστημα διασυνοριακών μικρών διαφορών γιατί δεν είναι επικίνδυνο θα έλεγα για τη εθνικά συστήματα. Ακριβώς γιατί αφορά διασυνοριακές διαφορές τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση για τις διασυνοριακές αυτές διαφορές, οπότε ο κόσμος αποθαρρύνεται και τις ε, αφήνει να περνάνε έτσι τώρα. Για τις ε, διαφορές κάτω από 12.000 ευρώ πράγματι υπάρχει ένα σύστημα, δεν είναι γνωστό και θα πρέπει άρα να υπάρξει ε, μεγαλύτερη διάδοσή του και διαφήμιση του θα έλεγα. Τώρα για το κατόφλι αυτό των 10.000 ε, ευρώ είμαι θα έλεγα θετικός και νομίζω πως ε, ούτως ή άλλως το σύστημα το οποίο υπάρχει δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι περισσότερο ένα είδος πειραματισμού. Αντιθέτως είμαι αντίθετος με την ιδέα που ακούστηκε από πολλούς ε, συναδέλφους για να γίνει διάκριση μεταξύ φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων. Είναι κακή η ιδέα, εγώ συμφωνώ με την εισηγήτρια εδώ πέρα. Δεν ε, υπάρχει θέμα απλοποίησης, αρκεί να γνωρίσει ο κόσμος το σύστημα και δεν χρειάζεται καμία άλλη διάκριση. Τώρα, ο βασικός λόγος για τον οποίο είμαι υπέρ του θέματος αυτού, ξέρετε πως δεν είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, είμαι υπέρ μιας Ευρώπης των Εθνών. Αλλά και σε αυτή την Ευρώπη των Εθνών θα υπάρχουν πάντα τέτοιες ε, διασυνοριακές ε, μικροδιαφορές, οπότε καλό είναι να έχουμε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ, έχετε τον λόγο. Για τις τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν στην πρόταση της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών, να προωθήσουμε δηλαδή το σύστημα ώστε να γνωρίζουν την ύπαρξή του. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να υποβάλουμε και εμείς παρόμοια σύσταση. Ακούστηκαν πολύ καλές ιδέες. Πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Όσον αφορά το όριο, η διαδικασία αυτή αφορά μόνο διασυνοριακές διαδικασίες. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί διαδικασία όταν μιλάμε για δύο άτομα που βρίσκονται στην ίδια νομική τάξη, στο ίδιο νομικό σύστημα. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε μέρη από διαφορετικά κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να χειριστούμε έτσι εγχώριες υποθέσεις. Εκεί εφαρμόζονται άλλες διαδικασίες. Πώς θα λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα στο μέλλον. Θα πρέπει να φροντίσουμε το σύστημα αυτό να μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο διαφόρων συστημάτων. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά, κάποιο από τη Λετωνία με κάποιον από το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε σαφώς οι αναλογίες είναι διαφορετικές. Η οικονομία της Πολωνίας, της χώρας μου, έχει αναπτυχθεί με απίστευτους ρυθμούς. Και οι τιμές είναι πολύ υψηλέ σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το όριο των 10.000 ευρώ. Αλλά Εάν δεν μα αρέσει ο όρος μικροδιαφορές, τότε μπορούμε να πούμε ε, διαδικασία για την επίλυση διαφορών μέχρι 12.000 ευρώ. Και όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα. Φυσικά θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την ύπαρξη του συστήματος, αλλά θέλουμε βέβαια να αποφεύγουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και ο κόσμος, ειδικά όταν συμμετέχει σε συναλλαγές στο διαδίκτυο, θα πρέπει να προσέχει. Όσον αφορά τη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ρυθμίσει αναλυτικά κάθε βήμα της διαδικασίας. Είναι επίσης χρήσιμο που αναφέρεται τι δεν καλύπτεται. Δεν έχω υποβάλει λοιπόν σχετική τροπολογία. Όσον αφορά τις υποθέσεις που βρίσκονται κάτω από το όριο, είναι σαφές ότι εφαρμόζονται άλλες διαδικασίες. Είναι σαφές πιστεύω το κείμενο. Μία πρόταση από μένα προς εσάς θα πρέπει να επιδιώξουμε την επίτευξη κάποιων συμβιβασμών. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε στο πλαίσιο των σκιωδών εισηγητών. Δεν ε, θέλω να συμπεριλάβω στο έγγραφο πράγματα τα οποία είναι ήδη προφανή. Θέλω το κείμενο να είναι απόλυτα απλό και σαφές. Και γι' αυτό είμαι υπέρ και ενδεχόμενων διαγραφών. Θα προετοιμάσω το έγγραφο και ελπίζω να το υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στο θέμα υπαριθμών 24. Και δίνω το λόγο στον κύριο Καβαντά. Ε, ευχαριστώ κάτι επί της διαδικασίας θα έλεγα. Δεν γνώριζα πως η Επιτροπή μας θα γίνει χώρος πειραματισμού για την ε, ψήξη του κλίματος. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τις υπηρεσίες ε, να τους ε, τονίσω πως ε, υποφέρουμε. Δεν είμαστε πολικοί οργανισμοί. Τραβάει το ρεύμα. Άλλοι συνάδελφοι έχουν βάλει τα παλτά τους. Σας παρακαλώ λοιπόν λύστε το να τελειώνουμε να έχουμε μια θερμοκρασία που θα μας βολεύει όλους. Ε, δεν είναι ανάγκη να πλευριτώσουμε τώρα. Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur Cavada, mais quand même la parole. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει παρόλα αυτά ο κύριος ε, Κοφεράτη, κύριε Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ζεστάνω εγώ το κλίμα λοιπόν, με τα λόγια μου. Κοιτάξτε, είχαμε νομίζω ήδη την ευκαιρία στην Επιτροπή μας να συζητήσουμε την ε, οδηγία αυτή και βεβαίως να ε, κάνουμε και την ακρόαση. Πριν τα Χριστούγεννα αυτό σήμερα έχουμε ένα άλλο βήμα θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με βάση τα έγγραφα που σας έστειλα με προτάσεις ε, με αλλαγές στις προτάσεις ε, τις αρχικές. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να συνοψίσω λίγο τα κεφάλαια στα οποία πρέπει να εστιάσουμε αυτά τουλάχιστον τα οποία θεωρώ εγώ τα βασικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε το δικαίωμα ταυτοποίησης των μετόχων ε, και την ε, διευκόλυνση ε, μετάδοσης πληροφοριών σε διαμέσους για τις ψήφους ακριβώς των μετόχων. Μετά έχουμε διαφάνεια θεσμικών επενδυτών και διαχειριστών κεφαλαίων, διαφάνειας συμβούλους κατεξιοδότηση και στους ε, μισθούς ε, των διευθυντικών στελεχών. Τέλος, ε, έλεγχη των συναλλαγών από ιδιώτες. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν είναι να καταλήξουμε με την οδηγία αυτή για να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ενός ε, συνολικού πλαισίου. για την διακυβέρνηση των επιχειρήσεων που ξέρετε πως είναι μεγάλο ζήτημα και καλύπτει την εταιρική κοινωνική ευθύνη και βεβαίως ε, αυτό το οποίο ο Ζακ Ντελόρ ε, είχε ήδη αναφέρει από το 1994 Βεβαίως, εκτός από τους ε, μετόχους, ε, πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, παραδείγματος χάρη τους ε, καταναλωτές. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Θα ήθελα τώρα να προσθέσω κάποιες λεπτομέρειες στα κεφάλαια που ανέφερα. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Όπως είπα, έχω κάνει κάποιες προτάσεις για αλλαγές έτσι ώστε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων να γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων για να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η μετάδοση προσωπικών δεδομένων ακριβώς για προστασία της ε, προσωπικής ζωής. Τώρα, μετάδοση πληροφοριών στις επιτροπές. Ε, κοιτάξτε, αυτό αφορά πολλά διασυν, πολλές διασυνοριακές δραστηριότητες. Η εξάσκηση των δικαιώματος ψήφου των μετόχων πρέπει να είναι εγγυημένη. και αυτό ακριβώς ενίσχυσα τους τομείς εκείνους που αφορούν την παροχή πληροφοριών για τους μετόχους των εταιριών, ειδικά αν τη ζητάει κάποιος ενδιάμεσος και βεβαίως και οι χρεώσεις και οι προμήθειες που παίρνουν αυτές αυτή η ενδιάμεση πρέπει να είναι διαφανής. Οπότε όταν μιλάμε για μακροπρόθεσμους μετόχους πρέπει να προστατευτούν αυτοί ιδιαίτερα γιατί ο στόχος ακριβώς της οδηγίας είναι να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες να βλέπουν τα πράγματα πιο μακροπρόθεσμα. Αντί για αυτή την βραχυπρόθεσμη προσέγγιση που βλέπουμε τώρα. Τώρα, για την διαφάνεια θεσμικών επενδυτών και συμβούλων κατά τα κτλ. Πρέπει νομίζω να τηρηθούν οι φυστάμενοι κανόνες διαφάνεια στην πρόταση της Κομισιόν, ειδικά για θεσμικούς επενδυτές. Πρέπει νομίζω να εγγυηθούμε πως οι θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές ε, κεφαλαίων και οι σύμβουλοι θα τηρούν έναν κώδικα συμπεριφοράς. Τέλος έχουμε τον ε, μισθό, ναι. την ε, αμοιβή των διευθυντικών ε, στελεχών, κάτι το οποίο είναι επίσης σημαντικό για να υπάρχει σωστή διαχείριση των επιχειρήσεών μας που θα αφορά και θα εστιάζει στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με την ε, πολιτική αυτή των ε, αμοιβών. Πρέπει λοιπόν να ψηφίζουν οι διευθυντές και για την εφαρμογή των μέτρων επαλήθευσης όπου αυτό απαιτείται. Επίσης ε, βάλα κάποιες ε, αλλαγές για να γίνει ακριβώς πιο διαφανής και η πολιτική ανταγωνισμού. Μία δυνατότητα είναι οι εργαζόμενοι να αναπτύσσουν ε, τις απόψεις τους για την πολιτική αμοιβών της εταιρείας. Δεν πρέπει αυτό να είναι προνόμιο μόνο των μετόχων πρέπει να υπάρχει έλεγχος από τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Ε, ε η αμοιβή των στελεχών μπορεί να συμπεριλαμβάνει και ε, το δικαίωμα απόκτησης ε, μετοχών αλλά ακριβώς αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη διαχείριση της εταιρεία. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε κάτι προς την κατεύθυνση της διαφάνειας με έναν τρόπο που θα ενθαρρύνει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα ξεπεράσει τα προβλήματα και τους κινδύνους που υπάρχουν στην κερδοσκοπία θα έλεγα. Πρέπει λοιπόν επίσης ε, να δούμε όλες τις διαφορετικές καταστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση χωρίς να προξενήσουμε κάποια βλάβη, κάποια αντίφαση. Δεν πρέπει να δώσουν υπερβολική δύναμη στους ε, μετόχους. Πρέπει να προσέχουμε ποιος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει στις γενικές συνελεύσεις. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά και σε προηγούμενες ε, συζητήσεις, γι' αυτό αναμένω να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων, ξεκινώντας με τους κοιόδης συζητητές και με όσους συμφώνησαν να υποβάλουν ε, τροπολογίες για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να υπάρχει μια ισορροπημένη και αποτελεσματική λύση. Τέλος, για το σημαντικό αντικείμενο αυτής της οδηγίας να ενισχύσουμε την ε, οδηγία μέσω των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό ακριβώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πράξεις κάτω εξουσιοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα μας και θεωρώ πως πρέπει να αποτελέσει τμήμα μιας εταιρική διακυβέρνησης προσανατολισμένης προς το μέλλον όπου θα καθορίζεται ο ρόλος του καθενός και τα πάντα θα είναι ισορροπημένα. Τέλος για το χρονοδιάγραμμα επειδή έγινε μια ερώτηση αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ε, προθεσμία για τροπολογίες. Έχει πάει τώρα στις 5 Φεβρουαρίου. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά θα έχετε λίγο χρόνο παραπάνω να το σκεφτείτε και να καταλήξετε σε κάποιες πιο προσεκτικές προτάσεις. Όπως είπα λοιπόν, Έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα, έχουμε λίγες μέρες παραπάνω για να κάνουμε έτσι λίγο καλύτερη δουλειά, αλλά ταυτόχρονα θα τηρήσουμε το πρόγραμμά μας. 5 Φεβρουαρίου λοιπόν τροπολογίες. ή 24 του σε εξέταση των ε, τροπολογιών και ψηφοφορία στην Επιτροπή ίσως μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αυτά από μένα. Αναμένω την άποψή σας και προτάσεις για τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε λιγάκι καθυστερήσει και στις 11.30 θα δεχτούμε τον Λετωνό Υπουργό Δικαιοσύνης. Ίσως λοιπόν να βιαστούμε λιγάκι, η συζήτηση να είναι πιο επικεντρωμένη στα ουσιώδη. Η Κομισιόν τώρα, κυρία Ιωάννα Σικούρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κοφεράτη για την εξαιρετική του έκθεση επί της προτάσεώς μας και είμαστε ευγνώμονες στον εισηγητή για την υποστήριξη του αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας που στοχεύει σε περισσότερο μακροπρόθεσμη, σε πιο μακροπρόθεσμη ε, επιχειρησιακή διακυβέρνηση. Πολλές ιδέες στην έκθεση αυτή είναι χρήσιμες και θα συμπλήρωναν πολύ καλά τις προτάσεις μας. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στην Κομισιόν καμιά φορά είναι δύσκολες οι συζητήσεις. Ε, μερικά θέματα δυσκολεύουν ιδιαίτερα τις χώρες μέλη και στο Συμβούλιο συνήθως μειώνεται, μειώνονται οι φιλοδοξίες μας για να υπάρξει συμβιβασμός. Γι' αυτό θεωρούμε σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και κάποια ευελιξία για να επιτευχθούν συμβιβασμοί. Δύο θέματα θα ήθελα να τονίσω. Ακούσαμε ιδέες για μεγαλύτερη εμπλοκή των ε, ενδιαφερομένων ιδιαίτερα των εργαζομένων. Εμείς δεν θα θέλαμε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο να υπερτονίσει το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων. Ξέρουμε ότι είναι λεπτό θέμα για τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι είναι σημαντικό το θέμα. και δεν αφορά μόνο τους μετόχους αλλά και άλλα τμήματα της, του δικαίου των επιχειρήσεων. Άρα ίσως να πρέπει να υπάρχει μια πιο ευρεία, πιο οριζόντια συζήτηση μεταξύ κομισιών ενδιαφερομένων κοινοβουλίου κρατών μελών. Αυτό προτείνουμε, να μην περιοριστούμε μόνο, να μην περιορίσουμε το εύρος των συζητήσεων. Όσο για την πρόταση να υπάρξουν πρόσθετοι μηχανισμοί, για την περισσότερη εμπλοκή των ενδιαφερομένων, να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα δηλαδή. Το βλέπουμε θετικά, αλλά πρέπει επίσης να εξετάσουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι εναλλακτικοί μηχανισμοί, γιατί μπορεί μερικοί να έχουν απρόβλεπτες ε, επιπτώσεις. Σε μερικά κράτη-μέλη έχει εφαρμοστεί το δικαίωμα της διπλής ψηφοφορίας, αλλά σε άλλα ή υπήρξε αρνητικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να τα ξανασκεφτούμε, να αξιολογήσουμε όλους τους μηχανισμούς για να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι. Τονίζουμε λοιπόν ότι θα δούμε το θέμα των κινήτρων για τους πιο μακροπρόθεσμα ενδιαφερόμενους ή μετόχους για να δούμε πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν κίνητρα για πιο υπεύθυνες επενδύσεις. Θα κάνουμε μία δημόσια διαβούλευση από την Άνοιξη ή και πριν. Και μετά θα προκύψει μια έκθεση που θα τα εξετάζει όλα αυτά βαθέως. Θα δούμε λοιπόν αυτό το θέμα των κινήτρων. Για να συνοψίσω λοιπόν, γνωρίζουμε ότι στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, συζητιέται επίσης το θέμα. Έχουμε δει μερικές από τις τροπολογίες τους. Με μερικές δεν συμφωνούμε και θα θέλαμε επίσης να πληροφορηθούμε για τις δικές σας τροπολογίες και ευχαρίστως να τις συζητήσουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας και σας κατευχαριστούμε κύριε Κομφεράτη. Ευχαριστούμε. Κυρία Βίξτρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάλι που βρίσκομαι εδώ στην Γιούρη και που ξανασυναντώ παλιούς και νέους φίλους. Όσον αφορά το θέμα αυτό, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του πάνω στο θέμα αυτό. Να τον ευχαριστήσω και για την πραγματική του προσπάθεια να ξυπνήσει το ενδιαφέρον μας ε, και τα έχει καταφέρει. Προσπάθησα να εξετάσω τις προτάσεις, αλλά πρέπει να εξετάσω κάποιες λεπτομέρειες και να συναντηθώ με ενδιαφερομένους ε, προτού να λάβω οριστική θέση. Αλλά ε, έχω κάποιες ιδέες τώρα. Η στόχη της Κομισιόν είναι πολύ καλή. Μ' αρέσει η ιδέα του να κινητοποιήσουμε την ε, μακροπρόθεσμη συμμετοχή των μετόχων στις εταιρείες ε, και να προωθήσουμε την διαφάνεια. Δεν αμφισβητώ τους στόχους, αλλά πρέπει να εξετάσουμε πιο αναλυτικά τον τρόπο επίτευξης των στόχων. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση. Εάν πρόκειτο να ψηφίσω την πρόταση της Κομισιόν όπως υποβλήθηκε σε εμά, θα πρέπει να ομολογήσω ότι δυστυχώς θα έπρεπε να συστήσω στην πολιτική μου ομάδα να την απορρίψει. Του, του λεχθέντος, ο μόνος τρόπος να προοδεύσουμε είναι να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση για να βελτιώσουμε την πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν. Νομίζω ότι με πολύ σκληρή δουλειά θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία να μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αλλά όπως είπα αυτό συνεπάγεται σημαντική αναδιατύπωση. Γενικά δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτό που χρειάζονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι υπερβολικά αναλυτικοί κανόνες από τους νομοθέτες τους. Μάλλον ήδη έχουμε υπερβολικά αναλυτικούς κανόνες. Επίσης δεν είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να δώσουμε κίνητρα για τη συμμετοχή των μετόχων ζητώντας από τις επιχειρήσεις να συντάσσουν αναλυτικά έγγραφα πολιτικής. Νομίζω ότι κινδυνεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε, να προσθέσουμε δηλαδή, να επιβάλλουμε πολύ γραφειοκρατία. σε ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες ήδη φέρουν πολλά βάρη. Και πράγματι η μακροπρόθεσμη συμμετοχή των μετόχων προέρχεται από την επιθυμία μας να βελτιώσουμε τις εταιρείες, αλλά δεν συνδέεται με την ανάγκη να εκπονούνται αναλυτικά έγγραφα πολιτικής. Με γνωρίζετε, είμαι φεντεραλίστρια, μ' αρέσουν οι πανευρωπαϊκές λύσεις. Νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις εξυπηρετούμε καλύτερα τις επιχειρήσεις με έναν ενίο ευρωπαϊκό νόμο αντί για 28 διαφορετικούς εθνικούς νόμους. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω το λόγο που έχουν υποβληθεί πολλές από τις προτάσεις σε αυτό το νομοθετικό πακέτο. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αμοιβή των διευθυντών, πιστεύω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του λέγειν των μετόχων όσον αφορά την αμοιβή, αλλά γιατί να υπαγορέσουμε μια τόσο αναλυτική ρύθμιση για το πώς θα γίνει αυτό. Ποια είναι η πραγματική μας ανάγκη εδώ. Λαϊκιστές όλων των ε, πολιτικών κατευθύνσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το θέμα της αμοιβή των διευθυντών για να συγκεντρώσουν περισσότερες ψήφους, αλλά μπορεί κανείς πραγματικά να ισχυριστεί ότι η απόδοση των ευρωπαϊκών εταιριών στην παγκόσμια οικονομία θα εξαρτηθεί από κάποιες μικρές ρυθμίσεις στην αμοιβή των διευθυντών. Σίγουρα όχι. Σημαντικό είναι τι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις να έχουν το χρόνο να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους αντί να ασχολούνται με την πλήρωση υποχρεώσεων που τους έχουν υποβάλει οι υπερβολικά φιλόδοξοι πολιτικοί και γραφειοκράτες της Ευρώπης. Οι μετοχοί θα πρέπει να ενδιαφερθούν για πράγματα πολύ πιο σημαντικά από συμβολικά θέματα όπως είναι η αμοιβή των διευθυντών. Σημαντική είναι η ταυτοποίηση των μετόχων. Νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να φέρει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως σε αυτό το σημείο του κειμένου είναι χρήσιμο να επικεντρωθούμε. Επίσης, όσον αφορά τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, με ανησυχεί η υπερβολικά αναλυτική ρύθμιση που υπέβαλε η Κομισιόν. Είμαι βέβαιη ότι εμπνεύστηκε από μια ευγενή βούληση να προστατεύσει τους μικρομετόχους, αλλά κινδυνεύουμε να επιβάλλουμε δυσανάλογα βάρη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κάτι που θα βλάψει την οικονομία μας και θα εξαλείψει τις προοπτικές για ανάπτυξη. Συνάδελφοι, θα ήθελα πολύ να μπορώ να είμαι πιο θετική, αλλά υπόσχομαι ότι θα εργαστώ επικοδομητικά με στόχο τη βελτίωση της πρότασης. Κύριε Κοφεράτη, Ειλικρινά δεν σας ζηλεύω που είσαστε εισηγητής για το περίπλοκο αυτό θέμα. Είμαι πεπισμένη όμως ότι θα μπορέσετε να συνδυάσετε τις διάφορες απόψεις ώστε στο τέλος να έχουμε μία πρόταση που να αντικατοπτρίζει τις θέσεις όλων και που να μπορέσει να συγκεντρώσει την υποστήριξη ευρείας πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Προσλέπω στην καλή συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πέντε ομιλητές και έχουμε δέκα λεπτά. Παρακαλώ να το έχετε κατά νου αυτό η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που υπέβαλε την πρόταση και που έχουμε τη δυνατότητα να τη συζητήσουμε τώρα εδώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα είμαι σύντομη. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τα προβλήματα από την οπτική της χώρας μου καθώς και τα προβλήματα που έχω με το σχέδιο έκθεσης και με την πρόταση της ε, Κομισιόν. Έχουμε ε, πάνω από 500 εισηγμένες εταιρείες, το 60% των ε, επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν δηλαδή ένα ή δύο μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και σε πολλές άλλες χώρες το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χθες και σήμερα, αργότερα σήμερα, θα ε, συζητήσαμε και θα συζητήσουμε το θέμα των ε, διοικητικών ε, συμβουλίων και της διαφάνειας. Όσο περισσότερη γραφειοκρατία, τόσο μεγαλύτερο βάρος επιβάλλουμε στις επιχειρήσεις. Θέλουμε διαφάνεια λοιπόν. Νομίζω ότι με την έκθεση του κυρίου Κοφεράτη επιβάλλουμε περισσότερη γραφειοκρατία αντί να απλοποιούμε τη διαδικασία. Επίσης, και στην έκθεση και στην πρόταση της Επιτροπής βλέπω να μην αναγνωρίζετε καθόλου το διτό σύστημα που έχει η Γερμανία. Έχουμε όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους, έχουμε και το Εποπτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο όργανο που συμμετέχει στις αποφάσεις της επιχείρησης. Με αυτά τα τρία σώματα, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, του Μετόχους και το Εποπτικό Συμβούλιο, έχουμε κατανομή των διαφόρων ρόλων. Η Κομισιόν αλλάζει τελείως την ισορροπία αυτή. Και το σύστημά μας δεν έχει λειτουργήσει καθόλου άσχημα τις τελευταίες δεκαετίες. Θα υποβάλω λοιπόν τροπολογίες όπου να δίνουμε βάρος στη διάκριση αυτού του ενιαίου συστήματος και του διτού συστήματος που έχουμε στην Γερμανία. Αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζεται και στο θέμα των αμοιβών των διευθυντών. Η αμοιβή των διευθυντών λαμβάνεται από τα συμβούλια αυτά. Γιατί λοιπόν να το αναθέσουμε αυτό αποκλειστικά στους μετόχους. Επίσης, όσον αφορά τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, πώς θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Κάθε φορά θα πρέπει να γίνεται συνέλευση των μετόχων. Αυτό στοιχίζει και καθυστερεί τις διαδικασίες σε μια επιχείρηση. Δεν είναι λοιπόν εφαρμόσιμες οι προτάσεις. Όπως και η συνάδελφος Βίκστρομ, βλέπω και εγώ επικριτικά την πρόταση. Αγαπητέ κύριε Κοφεράτη, ούτε κι εγώ σας ζηλεύω, είναι δύσκολο το έργο σας. Θα υποβάλω τροπολογίες και προσλέπω στην περαιτέρω ε, ε, αναλυτική συζήτηση της πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ καταλαβαίνω τις προθέσεις της πρότασης αυτής, αλλά δεν συμφωνώ όσον αφορά τις λεπτομέρειες. Μάλιστα θα ήμουν και πιο αγενής από τις ε, προλαλήσασες. Νομίζω ότι οφείλονται στην Κομισιόν πολλά προβλήματα. Όπως είπε και η συνάδελφος Νίμπλερ, έχουμε εδώ διάφορα σημεία. Τι γίνεται όσον αφορά τα επιχειρηματικά μυστικά. Θέλουμε σύστημα γρήγορο και ανταγωνιστικό. Εάν όλα θα πρέπει να συζητώνται στη συνέλευση των μετόχων, αυτό στοιχίζει χρόνο και χρήμα. Όσον αφορά την συναπόφαση των εργαζομένων. Και αυτό θα πρέπει να συζητιέται στη Γενική Συνέλευση. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα ο κάθε μέτοχος δεν ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα, επιστεύεται τη διεύθυνση. Επίσης, αναφέρθηκε το διτό σύστημα. Ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, των κρατών μελών, τα διάφορα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε αυτά και μήπως θα πρέπει να έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξης. Ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 3α έως δ, θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Αναφέρονται εδώ οι υποχρεώσεις ενημέρωσης. Δεν γίνεται εδώ διάκριση ανάμεσα στις μετοχές των ιδιοκτητών και στις ονομαστικές μετοχές. Στο 3 δ θα πρέπει να γίνει διάκριση. Μάλλον θα πρέπει να αναφέρεται ποιος πληρώνει. Θα πρέπει να διασαφινιστούν τα στοιχεία αυτά. Έχω διάφορες παρατηρήσεις, θα είμαι όμως σύντομος. Σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το θέμα της ευθύνης. Πέρα από το θέμα των δαπανών, ποιο πληρώνει δηλαδή. Σε περιπτώσει προβλημάτων θα πρέπει να είναι σαφέ ποιο είναι αρμόδιος, ποιο ευθύνεται για τι πληροφορίε αυτέ. Και επίσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών επιχειρήσεων υπάρχει το θέμα το γλωσσικό. Καταλαβαίνει κανείς όταν μιλάει η διεύθυνση στους μετόχους είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε αναλυτικά. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα σωστό δρόμο. Είμαι πάντως ιδιαίτερα επικριτικός όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ κύριο Σιέτσικα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης Αλλά ο άλλος κοιόδης του ΕΛΚ δεν είναι παρόν και μου ζήτησε να του παρουσιάσω τις, τα σχόλιά του. Τα περισσότερα τα είπε και η Αγγέλικα, η Σεσίλια ή ο Άξελ. Γι' αυτό δεν θα επαναλάβω τα ίδια, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο πράγματι. Ιδού τι φρονούμε ως προς την πρόταση της Κομισιόν και την έκθεση. Ο κύριος Κοφεράτη είναι συνάδελφος που τον εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά εμείς επικρίνουμε την πρόταση του. Γιατί θα είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή αν θέλουμε να λειτουργήσουν σωστά οι επιχειρήσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος πρόσθετης γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τελικά είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί κανείς να ανακατέψει εξαιρετικές ιδέες με πολύ άσκημες. Αν τα ανακατέψουμε όλα, τη συμμετοχή των μετόχων, των εργαζομένων κτλ, και μαζί με αυτά βάλουμε το ότι στις προσθήκες υπάρχουν και θέματα δικαιωμάτων ψήφου ή πλήρης ψήφου. Όλα αυτά είναι λάθος να τα ανακατέψουμε και να τα βάλουμε όλα μαζί. Πρέπει μάλλον να υπάρξει μια έκθεση για την πολιτική ευθύνη, περισσότερη ευθύνη των μετόχων. Αυτό ναι, αλλά όχι με πρόσθετες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις ο κ. μίλησε για το διπλό σύστημα της λειτουργίας των υποπτικών συμβουλίων. Αυτό υπάρχει και στη χώρα μου. Είναι όργανα που παίζουν κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν και οι μέτοχοι μετά που δίνουν εντολή στο όργανο αυτό για να παίρνει αποφάσεις. Αν κάτι δεν τους αρέσει μπορούν να υποβάλουν έτοιμα, να πούν αυτό και εκείνο δεν μου αρέσουν και θέλω να αλλάξει ούτως και Αντί να υπάρχει εδώ υποχρέωση κάθε τρία χρόνια να γίνεται μια νέα πολιτική και Και κάτι άλλο ακόμη, ξεχάσαμε μάλλον ότι εδώ μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικές στην ελεύθερη αγορά όπου ο καθορισμός των αμοιβών γίνεται ελεύθερα επίσης. Πρέπει αυτό να συνδέεται με το αποτέλεσμα της επιχείρησης, ναι λογικό θα ήταν, αλλά πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι κανόνες της αγοράς. Αν εμείς τώρα θέλουμε έτσι χοντροκομμένα και πολύ λίγο κομψά να επιβάλλουμε πράγματα που να αλλάξουν την κατάσταση σε ένα σύστημα που ήδη λειτουργεί, τότε εμποδίζουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων, δεν τη διευκολύνουμε. Θα καταθέσουμε πολλές τροπολογίες και ελπίζουμε τελικά να είναι αποδεκτό το σχέδιο έκθεση, αλλιώς θα το καταψηφίσουμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντουράν. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα, διότι μας ζητήσατε να είμαστε σύντομοι. Πρώτον, εγώ δεν επικρίνω καθόλου την έκθεση Κοφεράτη. Αντίθετα τον ευχαριστώ και τον συγχαίρω, διότι προσπάθησε στην έκθεσή του, και αυτό το δείχνει και η σημερινή συζήτηση, να αποδείξει ότι η οδηγία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί υπάρχουν στοιχεία και τάσεις που θα σκοτώσουν τελικά την επιχείρηση με την αυστηρά δημοσιονομική προσέγγιση. Οι επιχειρηματίες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να καταστρώσουν τη στρατηγική τους και όχι κοντόθωρα. Και πρέπει να καταλάβουν, όπως έκαναν και πριν, ότι είναι οι κύριοι παράγοντες της ανάπτυξης όχι μόνο δημοσιονομικά που είναι κοντόθερα πράγματα βραχυπρόθεσμα με μόνο στόχο το άμεσο κέρδος. Χρειάζεται μια λήψη υπόψη όντως των πραγματικοτήτων και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αλλιώς δεν θα επιβιώσει η ευρωπαϊκή οικονομία ούτε θα επανέλθει σε δυναμικότερα επίπεδα. Δεν είναι σωστό να αντι... φέρνουμε σε αντίθεση την γραφειοκρατία με την απαραίτητη απλοποίηση. γραφειοκρατία, είπαν μερικοί, ε, τρέφει το λαϊκισμό. Όχι. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι επενδύσεις και η μισθολογική πολιτική μπορούν να είναι παράγοντες ανάπτυξης. Πρέπει να ζητήσουμε περισσότερη διαφάνεια χωρίς να μιλάμε για παραπάνω γραφειοκρατία ως επίπτωση, αλλά να δούμε πώς ακριβώς γίνονται οι επενδύσεις στην Ευρώπη. Ας μην επανέλθω και εγώ σε πράγματα που είπαν άλλοι. Όλα όσα συμπεριέλαβε ο κύριος Κοφεράτη στην έκθεσή του για να ληφθεί εκ νέου υπόψη το μακροπρόθεσμος παράγοντας είναι όταν μου μιλάτε για γραφειοκρατία και μου λέτε ότι επιβάλλεται στις επιχειρήσεις πρόσθετα βάρη, μόνο κάποιος που δεν ξέρει την επιχείρηση, τις επιχειρήσεις τα λέει αυτά. Γιατί συνήθως στις ε, συνεδριάσεις των μετόχων όλοι ζητούν reporting για τους ε, επενδυτές και όχι ότι δεν συζητούν την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης γιατί η μεγαλύτερη υπεύθυνη για γραφειοκρατία δεν είναι οι βουλευτές, είναι οι δι... τυχοδιώκτες. Έπειτα, αφού μιλάμε για γραφειοκρατία, όλοι ξέρουμε τα κόλπα που γίνονται για τις επενδύσεις. Ώρες ολόκληρες προ προσπαθούν να κάνουν δημοσιονομική όπως λένε βελτιστοποίηση. Αυτό είναι γραφειοκρατία ή όχι. Και για να κάνουν αυτά τα κόλπα όλα χρειάζεται πολύ μεγάλη γραφειοκρατία πιστέψτε με. Αφού λοιπόν είμαστε στη μακροπρόθεσμη λογική και θέλουμε διαφάνεια πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση θα ωφεληθεί από τη διαφάνεια και θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία. Πρέπει να μπορούμε να γνωρίζουμε αναχώρα, δεν είναι δύσκολο, τον αριθμό των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, τους μισθούς και τους φόρους που πληρώνουν. Είναι πολύ απλό και θα επέτρεπε, μας επέτρεπε να γνωρίζουμε όταν έρχονται οι μέτοχοι να συζητήσουν, να γνωρίζουν και αυτοί που βρίσκονται τα κέρδη, ποια είναι ακριβώς τα έξοδα και τι γίνεται με τους φόρους. Πολύ σημαντικό για να βγούμε από την ε, βραχυπροθεσμική λογική και να μην σκεφτόμαστε μόνο την, το άμεσο κέρδος γιατί έτσι καταστρέφεται ολόκληρη η μακροπρόθεσμη στρατηγική των επιχειρήσεων. Όταν ο κύριος Γιούνκερ μιλάει για την ανάγκη των ε, περισσότερων επενδύσεων στην Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αγνοούμε ως ε, και αυτό πηγή κερδών. Κυρία Χάουταλα, μας περιμένει όμως απ' έξω ο ε, σύντομα. Ναι, ναι, σύντομα. Θα επικεντρωθώ στο άρθρο 9 γάμα. Γιατί το πρότυπο που προτείνεται εδώ χρειάζεται βελτίωση. Και η ανησυχία μας είναι ότι Εδώ καλύπτονται και δοσοληψίες της κανονικής καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αν αυτά θεωρηθούν related party transactions, τότε πράγματι θα επιβαρύνουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ελπίζω να το ξαναδούμε. Εγώ μιλάω για μια επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων που μπορεί να έχει χιλιάδες μετόχους και να χρησιμοποιεί πρώτες ύλες που αφορούν δοσοληψίες που ανέρχονται σε μεγάλο ποσοστό των δραστηριοτήτων της. Δεν πρέπει αυτές να τις καταστήσουμε αδύνατη τη λειτουργία τους. Μπορεί εκατοντάδες χιλιάδων τέτοιων δοσοληψιών να ενδιαφέρονται. Γι' αυτό να το ξαναδούμε, να μην κάνουμε την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων πιο δύσκολη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κοφεράτη, είναι σχεδόν αδύνατο αυτό που πρέπει να κάνετε. Πάρα πολύ σύντομα συμπεράσματα σας παρακαλώ. Ναι, πράγματι θα είμαι συντομότατος. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που μίλησαν για τις προτάσεις και συστάσεις τους καθώς και για τα σχόλιά τους που φαντάζομαι ότι θα τα μεταφράσουν σε τροπολογίες. Από ό,τι άκουσα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω τρία πράγματα. Πρώτον, ανταγωνιστικότητα και αγορά μια διευθετημένη αγορά είναι μια αποτελεσματική αγορά και ο οι κανονισμοί, οι κανόνες είναι χρήσιμοι. Όπου δεν υπάρχουν κανόνες συνήθως σημειώνεται αθέμητος ανταγωνισμός. Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα <clears throat> να πετύχουμε. Δεύτερον, η διαφάνεια. Όπου υπάρχει διαφάνεια υπάρχουν και πραγματικές σχέσεις, αλήθεια. Τρίτον, το μακροπρόθεσμα. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε συμπεριφορές που να μην είναι κοντόθωρες αλλά πιο μακροπρόθεσμες γιατί εκεί γίνονται οι επενδύσεις για να έχουμε κερδοφόρα αποτελέσματα. Περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία τις τροπολογίες σας. Σας είπα τις ημερομηνίες. 5 Φεβρουαρίου. Μετά θα τη συζητήσουμε 23-24 Φεβρουαρίου και θα εγκριθεί από την Επιτροπή μας 24 Μαρτίου. Ας προσπαθήσουμε να τα πετύχουμε αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Ευχαριστούμε πολύ κυρίε και κύριοι. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Το υπόλοιπο της πρωινής συνεδρίασης θα μεταφερθεί στο απόγευμα. μετά την προδιαγεγραμμένη συνεδρίαση του απογεύματος. Μετά θα συμπληρώσουμε με το υπόλοιπο του πρωινού. Η απογευματινή συνεδρίαση θα είναι συντομότερη από τη συνήθως, διότι το 34 πρέπει να αναβληθεί, επειδή ο εισηγητής είναι άρρωστος, ο κύριος Καρέμ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε την τιμή να καλωσορίζουμε τον εξοχότατο Υπουργό Ρας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 Ladies Κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ να προχωρήσουμε στο σημείο 29 της ημερήσιας διάταξής μας. Να καλωσορίσω θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Λετωνίας, τον κύριο Ράσνατς. Καλωσορίσατε. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Κάνει πολύ κρύο έξω. και περιμένουμε να ακούσουμε την ε, εισήγησή σας. Ε, θα αναφερθείτε στις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της λετωνικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης. Ακόμα μεγαλύτερη χαρά είναι να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας στη μητρική μου γλώσσα τα λετωνικά. Η Προεδρία θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τη Λετωνία, όχι μόνο επειδή είναι πρώτη φορά που θα προεδρεύσουμε στις εργασίες του Συμβουλίου, αλλά και επειδή αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Τα παιδεία αυτά είναι ιδιαίτερα επίκαιρα μετά από τα γεγονότα του Παρισιού. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να συλληπιθώ τους ανθρώπους της Γαλλίας για τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στο Παρίσι. Η Λετωνική Προεδρία καταδικάζει τέτοιες πράξεις ριζοσπαστικοποίησης. Θα πρέπει να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν στη Ρήγα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σε υπουργικό επίπεδο για μέτρα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει σοβαρά βήματα για να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και να μπορεί να συνεργάζεται πιο αποτελεσματικά για να προλάβει και να ερευνά τέτοια εγκλήματα. Γι' αυτό η Λετωνική Προεδρία θα θέσει τα θέματα αυτά, στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η πρόληψη και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει όχι μόνο τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, θα πρέπει όμως να βρει και τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε αυτό το θέμα και τις νομικές λύσεις που θα σέβονται τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ελευθερία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι επιτυχής και ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ελπίζουμε ότι ο τομέας της δικαιοσύνης θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Θέλουμε δηλαδή δικαιοσύνη για την ανάπτυξη. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης, ε, βασικό μου πεδίο είναι η δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Τα μέτρα στον τομέα της δικαιοσύνης συνδέονται όλο και πιο στενά με την οικονομική ανάπτυξη την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Τζούρι, σε θέματα αρμοδιότητάς της, θα ακολουθήσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2014. Θέλουμε λοιπόν δικαιοσύνη σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλουμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στα δικαστικά μας ε, συστήματα και θέλουμε να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η Επιτροπή Τζούρι δίνει βάρος στα θέματα αυτά, διότι ένα νομικά σταθερό περιβάλλον ένα νομικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ευημερία των ανθρώπων της Ευρώπης και είμαι βέβαιος ότι το καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με στενή συνεργασία ανάμεσα στους ε, τομείς δικαιοσύνης, ανάμεσα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης ε, και Εσωτερικών με την Επιτροπή Τζούρι. Τέσσερις βασικές προτεραιότητες λοιπόν έχουμε για τους επόμενους μήνες. Καταρχάς, θέλουμε να οροστικοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση που αφορά τα εμπορικό σήματα. Δεύτερον, θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο όσον αφορά την ε, ε, εξάλληψη της υποχρέωσης για την επικύρωση εγγράφων. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την πρόταση για τις μικροδιαφορές και να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τέταρτον, να εφαρμόσουμε την μεταρρύθμιση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας επιτέθη σημαντική συμφωνία κατά τους τρει τριμερεί διαλόγους που πραγματοποιήθηκαν. Δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας αυτή τη μεταρρύθμιση. Για να το πετύχουμε αυτό, με τη δική σας ε, συνεργασία θέλουμε να αφοσιωθούμε σε τεχνικά ζητήματα για να εντοπίσουμε τις εκκρεμότητες οι οποίες θα πρέπει να επιληθούν κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων. Θέλουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της Άνοιξης. Επίσης, θέλουμε να συζητήσουμε την οδηγία για τα επιχειρηματικά μυστικά και θέλουμε να την συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεύτερον, κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης δημοσίων εγγράφων ώστε να διευκολύνουμε την κινητικότητα των ανθρώπων. Η Λετωνική Προεδρία θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Μετά από μακροσκελή συζητήσεις στο Συμβούλιο, θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας πάνω σε αυτήν την νομική πράξη που θα επιφέρει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα από τα θέματα που εμπόδισαν την πρόοδο ήταν η διάσταση απόψεων σχετικά με το για ποια έγγραφα θα πρέπει να ισχύει η κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης. Τον Δεκέμβριο του 2014 το Συμβούλιο ΔΕΗ συμφώνησε πάνω σε μία ε, προσέγγιση που να βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης. Να ισχύει αυτό για ε, έγγραφα ληξιαρχικά. Θέλουμε να διευρύνουμε όμως το φάσμα των εγγράφων που θα καλύπτεται για να αυξήσουμε την ε, εμπιστοσύνη στα συστήματά μας. Θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε συμβουλία στο Συμβούλιο όσο γίνεται πιο σύντομα. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό τις σχετικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτον, κανονισμός για, τη διαδικασία, για την επίλυση μικροδιαφορών. Και εδώ το μέσο τη δικαιοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αποτελεί λοιπόν αυτό προτεραιότητα του θεματολογίου μας. Το Συμβούλιο ΔΕΗ κατέληξε σε θέση τον Δεκέμβριο του 2014. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας. Για να έχουμε καλή συνεργασία θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τα αποτελέσματα όλων των συζητήσεων στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε. Τέταρτον. Κατά τη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο και μάλιστα σύντομα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου. Όπως γνωρίζετε, το Γενικό Δικαστήριο ήδη χρειάζεται περισσότερο δυναμικό για να μπορεί να ολοκληρώνει τις υποθέσεις εν χρόνο. Μέσα, μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που το δικαστήριο υπέβαλε την πρόταση για τη μεταρρύθμιση το 2011, Έκτοτε, ο αριθμό ε, των εκρεμών υποθέσεων στο δικαστήριο έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε κάποιες περιπτώσεις, επιχειρήσεις περιμένουν πάνω από τέσσερα χρόνια για την έκδοση μιας απόφασης. Συχνά στο διάστημα αυτό ε, έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία των εταιριών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Για πρώτη φορά το ΔΕΚ έχει λάβει προσφυγή λόγω καθυστέρησης έκδοσης απόφασης ε, και μάλιστα με την απέτηση αποζημίωσης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις στο Συμβούλιο, πιθανότατα να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Θέλουμε, προτείνουμε μάλλον αναθεώρηση του δυναμικού που ήδη έχει στη διάθεσή του το ΔΕΚ. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια και να ολοκληρωθεί το 2019. Στην πρώτη φάση θα δημιουργηθούν 12 νέες θέσεις δικαστών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει συμφωνήσει. Στη δεύτερη φάση θα έχουμε 7 πρόσθετες ε, θέσεις ε, δικαστών επειδή ε, θα υπάρξει συγχώνευση με το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Η πρόταση της Προεδρίας ήδη προβλέπει 25% μείωση σε σχέση με την αρχική πρόταση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κόστος αυτής της μεταρρύθμισης ανέρχεται στο 0,01% του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η μη εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης θα έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακροπρόθεσμα. Ήδη τώρα θα πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανταγωνιστικότητά της. Κατά τη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας πάνω στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Γενικού Δικαστηρίου και να ξεκινήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε συμφωνία όσον αφορά τη μεταρρύθμιση αυτή. Παράλληλα θα πρέπει τα κράτη-μέλη μεταξύ τους να συμφωνήσουν όσον αφορά την διαδικασία διορισμού αυτών των νέων δικαστών. Μπορεί να είναι δύσκολο το θέμα αυτό, ελπίζουμε όμως να το ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Αξιότιμοι βουλευτές, πέρα από αυτές τις προτεραιότητες, η Λετωνική Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες της πάνω στα θέματα που εκκρεμούν, όπως είναι η οδηγία για τα δικαιώματα μετόχων ή την πρόταση για την μονοπρόσωπη εταιρεία. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε συζητήσει σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και σε πολιτικό επίπεδο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μέτρα που θα είναι απαραίτητα για να προωθήσουμε περαιτέρω τα θέματα αυτά. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, πάνω στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητα ε, του Υπουργείου Πολιτισμού στη Λετωνία. Επίση, θα συνεχίσουμε τι εργασίε μα πάνω σε θέματα ισότητα των φύλων, που αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού Κοινωνική Πρόνοια τη Λετωνία. Αυτά είναι θέματα που επίπτουν στι αρμοδιότητε τη Επιτροπή Τζουρί. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω ότι η Λετωνική Προεδρία θα εργαστεί πάνω στα θέματα αυτά. Εκ μέρους ε, του Συμβουλίου ΔΕΗ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ευρωβουλευτές ε, για τις εργασίες πάνω για την, επιτυχή ολοκλήρωση της... του κανονισμού ε, για την αφαιρεγγιότητα που θα ολοκληρωθεί μετά την εξέτασή του από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Είναι σημαντικό να μπορούμε να βρίσκουμε γρήγορες λύσεις για να προωθούμε την ευρωπαϊκή συνεργασία. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι μία από τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας σε όλους τους τομείς και στη δικαιοσύνη είναι η πιο στενή συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Θα συμφωνήσετε, πιστεύω, ότι η ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα είναι πολύ πιο επιτυχής εάν οι γειτονές μας είναι δημοκρατικές χώρες και χώρες όπου επικρατεί το κράτος δικαίου. Προσλέπω στην επιτυχή συνεργασία μαζί σας κατά τη διάρκεια του προσεχούς εξαμήνου. Αξιότιμοι βουλευτές, η Λετωνική Προεδρία είναι διατεθειμένη να βρει συμβιβασμούς για να βρεθούν λύσεις σε θέματα σημαντικά για τους ανθρώπους της Ευρώπης. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε από κοινό να καταλήξουμε γρήγορα σε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Η συνεργασία της Επιτροπής Τζούρι με το Συμβούλιο είναι προϋπόθεση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Τώρα, με την άδειά σας, τα μέλη της Επιτροπής θα ήθελα να κάνουν κάποιες ερωτήσεις και αν συμφωνείτε θα ακούσουμε αρκετές ερωτήσεις μαζί και μετά μπορείτε να απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις μαζί. Ε, μια που είμαι πρόεδρος, να το εκμεταλλευτώ και να κάνω την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Είστε διατεθειμένος επί Προεδρία σας να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Σβιεύκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε για την δυνατότητα που έχουμε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας, αλλά και για την δυνατότητα που έχουμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Προεδρία της Λετωνίας. πέντε προτεραιότητες για τους πέντε μήνες. Καλό νούμερο. Νομίζω, αν τα οργανώσετε θα τα καταφέρετε. Βεβαίως, ε, μια φορά δημιουργείται η εντύπωση πως κάνει κανείς περισσότερα από όσα είναι αναγκαία. Βεβαίως μετά έχουμε και την καλή συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Αυτό μπορεί να οργανωθεί εύκολα, νομίζω είναι σχετικά σαφές. Αναφέρθηκε επίσης το θέμα της ε, διαδικασίας ε, χρεοκοπίας έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά επί Ιταλικής Προεδρίας Νομίζω λοιπόν πως θα μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. πιο συγκεκριμένο τώρα. Μιλήσατε για το 10 και την αναγκαία αλλαγή της είναι πιο αποτελεσματικό. Θα έχετε την στήριξή μας. Έχουμε πάει πολλές φορές βεβαίως και στο Λουξεμβούργο να συναντήσουμε τους δικαστές. Θα μπορούσαμε να έχουμε και νέες ανταλλαγές ε, απόψεων, αλλά νομίζω πως όλοι συμφωνούμε στο εξής ε, πως ε, είναι ε, απολύτως απαραίτητη η ορθή λειτουργία και η μεταρρύθμιση του δικαστηρίου. Γιατί αν το αφήσουμε θα χειροτερεύσει η κατάσταση και μετά θα πάει πέντε χρόνια μια υπόθεση για να τελεσιδικήσει. Οπότε θα σας στηρίξουμε απολύτως. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς είναι το εξής. Έχετε κάποια πρόταση που θα μας επέτρεπε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Σταματά. Κύριε Υπουργέ, είναι ιδιαίτερη η στιγμή όπου έρχεστε ως πρόσωπος της χώρας σας 25 χρόνια μετά την απελευθέρωσή της να προεδρεύει την Ευρώπη. Και συμμερίζομαι και εγώ την υπερηφάνεια σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, αλλά πρέπει βέβαια να υπάρχει και αποτελεσματικότητα. Σας άκουσα, διότι την Προεδρία σας θα την ασκήσετε σε μια στιγμή όπου επανέρχονται γεωπολιτικά προβλήματα στην Ανατολή και επίσης σε μια στιγμή όπου η ανασφάλεια κυριαρχεί και πάλι στην Ευρώπη τρία κύματα τρομοκρατικών επιθέσεων τα τελευταία 25 χρόνια από τη Μαδρίτη μέχρι το Παρίσι. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι απλό. Πώς θα καταφέρετε να επωφεληθείτε με την καλή έννοια από τις συνθήκες αυτές για να διευκολύνετε τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Έχετε καμία πρόθεση λήψης μέτρων σε επίπεδο εισαγγελιών και συνεργασίας των, γιατί πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και το ίδιο γρήγοροι με τους εγκληματίες. Πρώτον ήταν αυτό. Δεύτερον και τελευταίον, δεν έχει γίνει καμία πρόοδος ως προς το σεβασμό της χάρτας των θεμελιωδών στην Ουγγαρία έχετε την πρόθεση να ασχοληθείτε και με αυτό. Γιατί γνωρίζετε ποιο θα είναι το τίμημα αν δεν γίνει τίποτα. Τέταρτο ερώτημα, Ράντιεφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την πρώτη σας ε, προεδρία και ελπίζω να μπορέσω να σας συγχαρώ και στο τέλος ε, της προεδρίας σας. Το ερώτημά μου είναι το ίδιο με αυτό που ακούστηκε πριν για τη Διοργανική Συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία που είναι μέλος ε, του προγράμματος εργασίας και πρέπει να συμφωνηθεί το συντομότερο δυνατόν για να έχουμε ακριβώς καλύτερη νομοθεσία. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς για να στηρίξετε την πρόταση της ε, Κομισιόν και να ε, προτρέψει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην συμφωνία αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις και μετά θα ακούσουμε άλλες τέσσερις εάν συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις αυτές ε, για τη διοργανική συνεργασία που αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές. Θα ξεκινήσω από εκεί. Να απαντήσω στην ερώτηση του Προέδρου και στην ερώτηση του κυρίου Ράντοφου. Βεβαίω η Προεδρία ενδιαφέρεται για την καλύτερη νομοθεσία και αναμένουμε καλύτερες προτάσεις και μια καλύτερη νομοθετική διαδικασία. Αλλά ένας από τους δείκτες πιο αποτελεσματικής τέτοιας διαδικασίας είναι το πόσο ε, ενεργητικά είναι τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, συμμετοχή τους στην διαδικασία αυτή. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι Υπουργοί να είναι πάντα παρόντες ε, και να εκπροσωπούνται οι χώρες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να συμμετέχουν και πιο ενεργά οι υπουργοί και με την ε, Κομισιόν και με τους ευρωβουλευτές των αντιστοίχων επιτροπών. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και παραμένει η η ίδια η δραστηριότητα λοιπόν η συμμετοχή των κρατών μελών των υπουργών είναι απολύτως αναγκαία όσον αφορά τώρα το 10 να ευχαριστήσω τον κύριο Σβιεύκα με, για τη δουλειά που έκανε για τον κανονισμό περί χρεοκοπίας και ως ένα βαθμό τον ζηλεύω γιατί σχεδόν τελείωσε και έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βεβαίως τώρα ξεκινάμε εμείς και το ερώτημα ήταν η μεταρρύθμιση του 10 και η διαδικασία αυτή. θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε από τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και την δυνατότητα να βρεθεί χρηματοδότηση. Ελπίζω όμως να καταφέρουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά τώρα τον διορισμό δικαστών και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, φαίνεται πως θα απαιτηθούν συζητήσεις γιατί οι απόψεις ε, ε, διαφέρουν όσο πιο εντατικά εργαστούμε, τόσο πιο γρήγορα βεβαίως θα βρούμε λύσεις. Αλλά θα δώσουμε οπωσδήποτε μια συγκεκριμένη λύση, πρόταση για λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Καβαντά μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ερώτησή σας. και πραγματικά είναι τιμή μας να προεδρεύουμε στο Συμβούλιο όπως είπατε και στις 25 χρόνια μετά την ανεξαρτησία μας. Όσον αφορά τα μέτρα τώρα για τις αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες, μαζί με το Συμβούλιο δικαιοσύνης ε, και εσωτερικών έχουμε προγραμματίσει ένα άτυπο συμβούλιο στη Ρήγα 19 και 20 Ιανουαρίου και νομίζω θα αποτελέσει μια σωστή βάση για την ε, περαιτέρω δουλειά μας. Έχουμε συμφωνήσει και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης ε, της Γαλλίας Έχω ακούσει πολλές ε, διαφορετικές ιδέες. Ακόμα και ιδέες ε, για δημιουργία ενός ευρωπαϊκού FBI ή κάτι τέτοιο. Αλλά βεβαίως γνωρίζω πως ε, πολλοί υπουργοί έχουν συγκεκριμένες προτάσεις και οπωσδήποτε το άτυπο συμβούλιο στη Ρήγα θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για το αστικό δίκαιο και το οικογενειακό δίκαιο πιο συγκεκριμένα. Χθες είχαμε την κυρία Γιούροβα εδώ πέρα και μας είπε πως ε, συνεχίζει να ασχολείται με κάποια θέματα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα τις συνέπειες ότι πολλά καρτιμέλη έχουν ήδη το Σύμφωνο Συμβίωσης Ατόμων ε, του Ιδίου Φύλου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια θα είναι η συνεισφορά της χώρας σας ε, στην Προεδρία σας και ίσως θα μπορούσατε να τονίσετε και κάποια άλλα πράγματα που θα είναι σημαντικά για εσάς στον τομέα του βαστικού δικαίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γκούταλαντ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να σας κάνω αυτή την ερώτηση εγώ είχα προσωπικά μελετήσει την ε, Λετωνία στη μεταβατική της περίοδο όταν ε, σπούδαζα και χαίρομαι που τώρα λαμβάνεται την εξουσία. Έχω όμως μία ερώτηση όσον αφορά τις θηγατρικές εταιρείες. για τις ε, ευρωπαϊκές αυτές ε, εταιρείε ε, και νομίζω πως συμφώνησε και μία συνάδελφος πως μπορούμε να οδηγηθούμε σε εταιρείε οι οποίες δεν είναι ακριβώς και πολύ σοβαρές και ανταυτού θα οδηγούνται σε εταιρείε οι οποίε θα διαλέγουν ακριβώ που θα προσφεύγουν. Δηλαδή, αν μπορούν να εγγράφονται σε ένα κράτο μέλο, να λειτουργούν σε άλλο μετά, δηλαδή να είναι ουσιαστικά γραμματοκιβώτια αντί για πραγματικές εταιρείε. Ένα πρόβλημα και φορολογικό οπωσδήποτε, αλλά και για τα συνδικάτα και για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οπότε, έμαθα ότι θα κάνετε σεμινάριο με εμπειρογνώμονες, αλλά θέλω να ακούσω και την άποψή σας εδώ πέρα. Γιατί με την πρόταση που έχουμε τώρα, ίσως οδηγηθούμε σε εταιρείε όχι μη σοβαρές, που θα ψάχνουν βεβαίως τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν θέλουμε. Θέλω λοιπόν την άποψή σας εδώ πέρα. Ευχαριστώ, κύριο Σάντερσον. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι καλή Προεδρία. Και εύχομαι η επιθυμία η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι μετά τα γεγονότα στο Παρίσι ελπίζω να μην οδηγήσει σε άσοφες κινήσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την σύμβαση του Μαρακές για τυφλούς και άλλους και την πρόσβαση σε έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει αυτήν την συνθήκη και πρόκειται να επικυρωθεί. Περιμένουμε λοιπόν εναγωνίως μήνυμα από το Συμβούλιο για να προχωρήσουμε. Υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει το θέμα στο Συμβούλιο. Ελπίζω όμως η Λετωνική Προεδρία να λύσει αυτό το θέμα πολύ σύντομα. Μήπως μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Thank you. Uh, Mrs. Ευχαριστώ κυρία Γκάρικα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό για την πολύ συγκεκριμένη απάντησή του στα ερωτήματα που τέθηκαν. Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ καλά αυτά τα νέα που μας δίνετε. Καλό είναι που έχετε ορισμένα σχέδια και προθέσεις όπως το θέμα με το οποίο ασχολούμε αυτή τη στιγμή και θα κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε χρήσιμους συμβιβασμού. Ένα άλλο αίτημα που έχω κύριε Υπουργέ μου στο Συμβούλιο θα προεδρεύσετε πολλές σημαντικ... πολλών σημαντικών συνεδριάσεων και με ενοχλεί το ότι σε δύο κράτη μελη η, χώρα, η χάρτης των θεμελιωδών δεν εφαρμόζεται όπως και στη χώρα μου. Συνήθως το ξεχνάμε. Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να υποφελούνται από την ίδια νομική προστασία. Αν έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να το πράξετε θα ήθελα να μου πείτε, να μου σχολιάσετε αυτό το θέμα να ζητήσετε δηλαδή από όλες τις χώρες να εγκρίνουν το έγγραφο για να δίνεται η προστασία σε όλους τους πολίτες όλων των χωρών. Ευχαριστούμε. Τελευταίο ερώτημα. Κύριος Μπουντά. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας ρωτήσω τι φρονείτε για την ανάγκη ευρωπαϊκής διευθέτησης του θέματος των χρεοκοπιών φυσικών προσώπων γιατί αυτή τη στιγμή αφορά μόνο τις εταιρείες, νομικά πρόσωπα δηλαδή. Γιατί, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να χρεοκοπήσουν. Ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει και σοβεί αυτή η οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Πολλές φορές οι τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια τους και τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν πια να αποπληρώσουν τις δόσεις τους. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ μου έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για, τα ερω... για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά με την οποία τέθηκαν. Αρχίζω λοιπόν με την κυρία Χάουταλα. Φυσικά τα θέματα που αναφέρατε είναι λεπτά. Λεπτά. Ιδιαίτερα εκείνα των διαμεθοριακών Πρέπει να πω ότι τα κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν αποκρισταλώσει την άποψή του Η Λετωνική Προεδρία με βάση τις ευχές των χωρών μελών δεν προτίθεται να οργανώσει πολιτική συζήτηση του θέματος. Προβλέπεται στο Συμβούλιο να συνεχιστούν οι συζητήσεις το δεύτερο ημίση, την άλλη Προεδρία του Λουξεμβούργου. Αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα για καταπολέμηση της άνησης μεταχείρισης και εννοώ οποιοδήποτε τύπου, τότε μπορώ να πω ότι κατά την Προεδρία μας θα την υποστηρίξουμε, θα υποστηρίξουμε τέτοιο αγώνα. Γιατί είμαστε κατά οποιασδήποτε άνησης μεταχείρισης σε όλα τα κράτη-μέλη. Αφού όμως μιλάμε για θέματα αστικού και οικογενειακού δικαίου υπάρχουν εδώ διαφορές μεταξύ χωρών μελών και δική τους δικαιοδοσία είναι να αποφασίσουν ποιες σχέσεις θα αναγνωρίσουν. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις και δικαστικές από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάθε φορά τα κράτη-μέλη λέγεται ότι πρέπει να αποφασίζουν. Ακόμη για το αστικό δίκαιο το θέμα της απαγωγής παιδών είναι και αυτό πολύπλοκο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών. Η επόμενη τεχνική ανάλογη συνεδρίαση είναι 28 Ιανουαρίου. Και βέβαια η περίπτωση 1.13 θέτει πρόσθετα ερωτήματα και προβλήματα. ως προς το πώς θα εφαρμοστεί μελλοντικά το εργαλείο αυτό. Επόμενο ερώτημα επόμενο. της κυρίας Γκούτλαντ. για τις εταιρείες μονομελούς προσωπικού. Η Ιταλική Προεδρία πέτυχε σημαντική πρόοδο γι' αυτό και εμείς θα προσπαθήσουμε απλώς να τελειώσουμε το θέμα ώστε να, λάβουμε, να δοθεί εντολή διαπραγματεύσεων από το Κοινοβούλιο. Όσο για την έδρα των επιχειρήσεων, και αυτό είναι επίκαιρο θέμα και από τα κυριότερα της πρότασης και θα αναζητήσουμε και από αυτού συμβιβασμό κύριος Άντερσον. Μίλησε για τη συμφωνία της Μαρακές. Η Λετωνική Προεδρία υποστηρίζει τη συμφωνία αυτή για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τυφλών και ανθρώπων με προβλήματα όρασης ώστε να απολαμβάνουν πλήρως τη ζωή και αυτή και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εγκριθεί στο όνομα ολόκληρης της Ένωσης αυτή η συμφωνία. Τώρα, για τον κύριο Γκέριγκερ, κύριο Ξέρουμε ότι η κύρωση της χάρτας είναι σημαντικό θέμα και το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ελπίζω να την, επικυρώσουν όλα τα κράτη-μέλη και τα υπόλοιπα δηλαδή. Ο κύριος Μπούντα μίλησε για τη χρεοκοπία φυσικών προσώπων. Ναι και αυτό είναι θέμα που συζητιέται και σε όλες τις χώρες μέλη και είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι το σκάσιμο της οικοδομικής φούσκας έπληξε πολλές χώρες πολύ σκληρά. Ολόκληρη γενιά σε μερικά κράτη-μέλη φέρει ακόμη το ένα επαχθές βάρος χρέους και οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα θα την υποστηρίζαμε. Σε πολλές χώρες μέλη η αρχή του ετοιμοπαραδότου εφαρμόζεται και πολλές φορές διαφοροποιεί το δίκαιο στις χρεοκοπίες φυσικών με νομικών προσώπων. για να μπορούν μέσα σε ένα χρόνο να υπολογίζονται οι πραγματικές ζημίες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των δανειστών, αλλά και το lobbying από εμπορικές τράπεζες. Όλα εξαρτώνται από το πόσο καλά θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Όσο για το νέο κανονισμό θα διευκολύνει τις διαδικασίες για διαμεθοριακά θέματα προφανώς. Κύριε Υπουργέ, έχουμε εξαντλήσει τις ερωτήσεις από τα μέλη. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας. Όπως βλέπετε η Επιτροπή μας είναι ανοιχτή σε συνεργασία με την Προεδρία σας και ειλικρινά ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να σας συγχαρούμε και στο τέλος της Προεδρίας. λόγω των επιτυχιών που θα έχετε καταρθώσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσέλευσή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια ακόμη ανακοίνωση. Για το σημείο 27 TTIP που πρέπει να το αναβάλουμε μέχρι την επόμενη μας συνεδρίαση γιατί ο κύριος Φώσο εισηγητής δεν μπορεί να προσέλθει το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. <coughs> Καλή όρεξη.